να τη βοηθήσουμε καλύτερα με άλλο τρόπο και να αφήσουμε την Ουκρανία σαν μια υπερήφανη ανεξάρτητη χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάμπελ Μπάνεμαν. Η κυρία Σέιντι έχει το λόγο. Ο κύριο Σέιντι. Ευχαριστώ